σε παράγραφος 2. Οι αρμόδιες επιτροπές ε, διαβίβασαν τρία διορθωτικά κείμενα στα κείμενα τα οποία εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βάσει του άρθρου 231 παράγραφος 4 του κανονισμού αυτές οι διορθώσεις εγκρίνονται εάν εντός 24 ώρων μετά από την ανακοίνωσή τους ε, δεν ε, ζητήσει να ε, ψηφιστούν. Οι διορθώσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας και οι τίτλοι τους θα δημοσιευτούν στα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.